στη φάση αυτή να περάσουμε ένα σαφές μήνυμα για το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε τόσο ώστε να πετύχουμε ένα πραγματικά ουσιαστικό και ουσιαστικό, ένα πραγματικό και ουσιαστικό στόχο εξοικονόμηση ενέργειας. Ευχαριστώ κύριε Μπένσεν, ευχαριστώ συνάδελφε, ευχαριστώ επίτροπε. Φτάνει τελείωσε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 και περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, στην επόμενη έκθεση. κατάργηση οδηγιών σχετικά με τη μετρολογία. Πρώτος ομιλητής, η κυρία Βάισγκέρμπερ. Θα περιμένω να, λάβουν τη θέση, να λάβει τη θέση του ο Επίτροπος. Η κυρία Weisgerber. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδες εισηγητές της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και όλους όσους συνέβαλαν σε αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα. Χωρίς ε, την επικοδομητική και ειλικρινή συνεργασία με την Επιτροπή και με την Βελγική Προεδρία δεν ε, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αυτό το δοσιέ. Όπως ε, μπορείτε να φανταστείτε, είμαι πολύ ευχαριστημένη ως ηγήτρια με αυτό το αποτέλεσμα. Γιατί θα υπάρξει κατάργηση, κατάργηση 8 οδηγιών που είναι παροχημένες και αυτό συνιστά ένα βρήμα προς την κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας στην Ευρώπη. Ενδιαφέρον σε αυτές τις οδηγίες είναι το γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό θεωρούνται παροχημένες γιατί έχουν αντικατασταθεί από διεθνείς κανόνες που ανταποκρίνονται στο επίπεδο της τεχνολογίας. Πολύ συχνά οι χώρες ε, πολύ συχνά είναι παροχημένες οι εθνικές νομοθεσίες. Εδώ θεωρείται παροχημένη η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εάν, αν θέλουμε να έχουμε ε, λιγότερη γραφειοκρατία μέχρι το 2012, θα πρέπει να, να πάρουμε ξεκάθαρα θέση. Για να... Και θα πρέπει, όπως είπε ο κ. Στόιμπερ, να αρχίσουμε να σφυρίζουμε δυνατά στην Ευρώπη, δηλαδή να προχωρήσουμε στην πράξη. Αλλά πολύ συχνά ο διάβολος αποκρύπτεται στις ε, λεπτομέρειες, όπως το δείχνουν αυτές οι οχτώ οδηγίες σε σχέση με την ε, μετρολογία οδηγία σχετικά με τις μετρητές ψυχρού ύδατος και τα κάθαρτα ύδατα, ε, σχετικά με, την, ε, με τα πιεσόμετρα και ελαστικά αυτοκινήτων οχημάτων ή σχετικά με τη μάζα εκατολίτρου των δημητριακών ή σχετικά με την καταμέτρηση της χωρητικότητας των δεξαμενών των πλωτών μέσων. Οι οδηγίες αυτές έχουν αντικατασταθεί από πιο... τα όργανα αυτά μέτρηση έχουν αντικατασταθεί από πιο σύγχρονα ψηφιακά όργανα και γι' αυτό μπορούν να καταργηθούν αυτές οι οδηγίες. Αυτό δεν έχει επιπτώσει στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ούτε στο υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών που είναι ιδιαίτερο σημαντικό για μα. Παρ' όλα αυτά, το συμβόλιο ε, έχει μπλοκάρει το θέμα αυτό για πολύ καιρό. Αλλά πετύχαμε στο πλαίσιο του τριμερού διαλόγου να βρούμε ένα λογικό συμβασμό και στην πρώτη ανάγνωση, κάτι που συνήθως είναι εξαίρεση μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Η οδηγία για την καταμέρηση ορκιότητα των δεξαμενών ε, θα καταργηθεί ε, στις 11 Ιουλίου του 2011 οι υπόλοιπες ε, οδηγίες θα καταργηθούν αργότερα. Μία νέα πρόταση θα υποβάλει η Κομισιόν τον Απρίλιο η βασική ιδέα είναι ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει ποια τμήματα των παλαιών οδηγιών θα πρέπει να διατηρηθούν και να ε, ενσωματωθούν ε, στη νέα οδηγία. Όπως ε, για παράδειγμα ε, στην οδηγία σχετικά με τα πιεσόμετρα εγκαλαστικά αυτοκινήτων. Ε, τα τμήματα αυτά, αν έρθουν, ε, λογικά αυτά τα στοιχεία, θα συμπεριληφθούν στη νέα οδηγία. Έτσι βλέπουμε λοιπόν ότι η Ευρώπη θέλει πράγματι να μειώσει τη γραφοκρατία και να δημιουργήσει προποθέσει για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Είμαι υπερήφανη για το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη δική του εισφορά για τη μείωση τη γραφειοκρατία και για την ε, ταχύτερη ε, εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Τώρα, θα ήθελα να πω κάτι για τους πίνακες ε, συσχετισμού συνάφειας. Είναι οι πίνακες που θα πρέπει να καταρτήσουν οι χώρες μέλη για να αποδείξουν πώς έχουν προβεί στην ε, εφαρμογή της οδηγίας. Εμείς έχουμε μια πιο ήπια, μια πιο ήπια διατύπωση αλλά παλέψαμε για μια πιο αυστηρή διατύπωση στο μέλλον. Και θεωρώ ότι και αυτή είναι μια επιτυχία που χρωστάμε στους ε, σκιώδεις ηγητές της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ταλιάν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κυρία Βάις Γκέρμπερ για το έργο, το διεξοδικό έργο που ανέλαβε για μια περίπλοκη σύνθετη πρόταση που είναι το αποτέλεσμα μια μακράς συζήτηση. Η δουλειά τη λοιπόν δεν ήταν εύκολη το γεγονό ότι επιτυχάνουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση σημαίνει ότι η συγκήτρια ήταν εξαιρετικά ικανή να πετύχει συμφωνία. Η απόφαση αυτή είναι μια σημαντική φάση για την απλοποίηση της, ε, νομοθετική, της έξυπνης ε, νομοθετικής ρύθμισης. Η better regulation πρέπει να γίνεται όλο ένα και περισσότερο ένα στόχος των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και, της Επιτροπή, και η Επιτροπή συμφωνεί απόλυτα ότι πρέπει να στοχεύει πάντα στην βελτίωση της κοινωτικής νομοθεσίας. Η πρόταση αυτή καταργεί οκτώ πεπαλαιωμένες οδηγίες για έξι κατηγορίες ε, ε, οργάνων μέτρησης, διότι τα μέτρα αυτά έχουν ξεπεραστεί και οι εμπορικές, ε, σχετικές εμπορικές ανταλλαγές μειώνονται. Επιπλέον δεν υπάρχουν εμπόδια για την ε, εμπορία υποκατάσταση των προϊόντων που είναι τεχνικά πιο εξελιγμένα στο πεδίο εφαρμογή τη οδηγία. Στο μέλλον τα κράτη-μέλη θα μπορούν να έχουν ε, εθνικά όργανα, αλλά τούτο δεν θα εμποδίσει τις ανταλλαγές, διότι υπάρχουν διεθνεί κανόνες που ήδη ρυθμίζουν πλήρως τα παλιά αυτά εργαλεία και την πλειοψηφία των προηγμένων ε, υποκατάστατων προϊόντων. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπόδιο έχει μια συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόδιο που επιβάλλει σε κάτι μέλη να βασίζουν την νομοθεσία του στι διεθνεί ε, αυτέ προδιαγραφέ. Η συνθήκη τη Ένωση επιβάλλει στα κράτη-μέλη την αναγνώριση ε, ισοδύναμων προϊόντων που είναι νόμιμα στο εμπόδιο σε ένα άλλο κράτο μέλο. Η Επιτροπή δέχεται λοιπόν θετικά τη συμβαστική πρόταση σε πρώτη ανάγνωση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου που προβλέπει την κατάργηση τη οδηγία τον Ιούλιο του 2011 και των άλλων 7 οδηγιών το Δεκέμβριο του 2015. Η Επιτροπή επίσης δηλώνει εκ νέου ότι είναι έτοιμη να εξετάσει τα επιχειρήματα υπέρ της εναρμόνισης που θα υποβληθούν, κάτι διάρκεια, που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Επίσης τονίζουμε ότι τα εργαλεία αυτά θα εξεταστούν μέχρι το τέλος του έτους και αν δούμε ότι χρειάζεται θα υποβάλουμε ε, σχετική νομοθεσία βάσει των αρχών του, ε, της έξυπνης νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Κύριε Κόμη, έχετε το λόγο. Υποστηρίζω απόλυτα την θέση της εισηγητρίας για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την κατάργηση οκτώ οδηγιών στον τομέα της μετρολογίας. Ιδίως δέχομαι θετικά την πρόταση για την παραχώρηση στα κρατημέλη επαρκούς χρόνου για την αξιολόγηση των πιθανών συνεπειών της κατάργησης στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας ομικρονόμικων ε, μη συμφωνώ με τους ε, στόχους ε, της, ε, του Better Regulation και την απλοποίηση που προωθεί η στρατηγική της Λισαβόνας μεταξύ άλλων. Θεωρώ ωστόσο ότι είναι σημαντικό να δώσουμε στα κράτη-μέλη επαρκή χρόνο για να εξετάσουν και να παληθεύσουν ότι η κατάργηση των οδηγιών αυτών δεν θα προκύψει μια νομική μια έλλειψη ασφαλεία δικαίου. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει να μειωθούν οι ανησυχίες που εκφράστηκαν από διάφορα κρατημέλη για την αδυναμία να έχουν επαρκή χρόνο για να αντιμετωπίσουν ε, την ε, νομοθετική, το νομοθετικό κοινό που θα δημιουργηθεί μετά την κατάργηση. Ε, Άρα βλέπουμε ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική συμβαστική λύση μεταξύ της θέσης επιτροπής που είναι υπέρ της πλήρους κατάργησης των οδηγιών και αντίθετη με τη νέα νομοθετική ρυθμίση του θέματος στο πλαίσιο της οδηγίας όμικρον μη και των αρχικά επικριτικών ε, θέσεων των κρατών μελών εν της προτάσεις αυτής. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ε, ε, ευχαριστούμε πολύ κυρία Βάζ Κέρμπερ για την καλή συνεργασία που είχαμε. Εξ ονόματος της ομάδας μου θα ήθελα να πω ότι εγώ δεν ε, διαπνέομαι από την ίδια εφορία όσον αφορά την κατάργηση αυτών των οχτώ οδηγιών. Γιατί πράγματι υπάρχουν ορισμένα πεπαπαλαιωμένα όργανα μέτρησης των οποίων οι ρυθμίσεις θα καταργηθούν αλλά στις συζητήσεις διαπιστώσαμε ότι όπως το είπατε και εσείς η ίδια ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και υπήρξαν πολλές δυσκολίες για να διαπιστώσουμε ποιος είναι πραγματικά ο δεδειγμένος δρόμος. Η πολιτική μου ομάδα θα υπερψηφίσει αυτό το συμβιβασμό γιατί είχαμε την διαβεβαίωση από την Κομισιόν ότι θα εξετάσει εφόσον παρήσατε η ανάγκη ε, την ε, συμπερίληψη αυτών των, κάποιων τμήματων των παλαιών οδηγιών στην όμικρον όμικρον μη. Και θεωρώ ότι αυτό θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη της Επιτροπής. Υπό την προπόθεση αυτή είπαμε ναι, θα υποψηφίσουμε το συμβιβασμό γνωρίζοντας ότι πράγματι θα πρέπει να εξεταστούν κάποια στοιχεία. Όσον αφορά τους πίνακες ε, συσχετισμού, θα ήθελα να πω ότι οι συνάφειες θα πρέπει να πω ότι είπαμε ότι αποδεχόμαστε αυτή την ήπια διατύπωση μεν, αλλά πράγματι αυτό είναι από τα τελευταία κείμενα που δεχόμαστε μια τέτοιου είδους ε, ήπια διατύπωση, γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό δίκαιο το οποίο έχει συμφωνηθεί από τις χώρες μέλη και το οποίο να εφαρμόζεται πράγματι με σωστό τρόπο. Αυτό όμως μπορούμε να το εξετάσουμε μόνο εφόσον έχουμε τις πληροφορίες και τις πληροφορίες θα τις αντιλήσουμε από αυτούς τους πίνακες συσχετισμού και βάσει των πινάκων αυτών θα κάνουμε τη σχετική ανάλυση. Ευχαριστώ κύριε Μπουσόη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή και τους ε, αδέλφους που συνέβαλαν στην προετοιμασία αυτής της έκθεσης φαινόταν ότι ήταν ιδιαίτερα τεχνικό το έργο αλλά ε, τελικά διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν λύσεις. Σκοπός να πλουστευθεί το κοινοτικό κεκτημένο καταργώντας οδηγίες που αναφέρονται σε όργανα μέτρης που χρησιμοποιούνται πλέον λόγω των διεθνών προτύπων και της προόδου της τεχνολογίας. Είναι λογική η προσέγγιση Επιτροπής. αν η αρχή της αναγνώρισης ισχύει ώστε να, ε, ε, να επιτρέπει την ελεύθερη ελεύθερη κυκλοφορία, δεν, νέα, δεν απαιτούνται περαιτέρω ρυθμίσει, και τεχνικές προδιαγραφές θα εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη. Η των οδηγιών δεν πρέπει να οδηγήσει σε νέους ε, εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία ή να προσθέσει βάρος στις εθνικές διοικήσεις. Δεν πρέπει να υπάρξουν κενά μεταξύ της κατάργησης των παλαιών οδηγιών και την θέσπιση της οδηγίας για τα όργανα μέτρησης. Η έκθεση στην ΙΜΚΟ προέβαλε, έλαβε υπόψη τη δυνατότητα να, καλυφθούν, να καταργηθούν οι, οι, τα, οδηγίες δίνοντα επαρκή χρόνο στη, στα κράτη-μέλη, ώστε μήπως δημιουργηθεί νομική αβεβαιότητα μετά την κατάργηση των οδηγιών αυτών. Τα, μέτρα, ε, τα όργανα μέτρηση, επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δει κατά πόσο ορισμένα από τα όργανα μέτρησης των οδηγιών που καταργούνται πρέπει να συμπεριληφθούν στην όμικρον όμικρον μη, την οδηγία για τα όργανα μέτρησης. Εγώ σας προτείνω να ε, ψηφίσουμε υπέρ της ε, έκθεσης στην πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την καλή συνεργασία με τους σκιώδεις. Θα είμαι σύντομη γιατί νομίζω ότι τέθηκαν όλα τα σημαντικά σημεία. Η πολιτική μας ομάδα βεβαίως θα υπερψηφίσει το συμβασμό αλλά θεωρούμε ότι η Κομισιόν ε, στην ε, αναθεώρηση ε, θα διατηρήσει μια κριτική ματιά και είμαστε ευτυχείς που βρήκαμε αυτό το συμβασμό όσον αφορά τους πίνακες συσχετισμού. Αλλά ο συμβασμός ε, έχει μια ημερομηνία λήξης ε, και το Συμβούλιο θα πρέπει να αντιδράσει ε, και εμείς δεν θα υποχωρήσουμε εδώ γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιδράσουν και οι χώρες μέλη. Ο κύριος Κοζούσνικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, προσωπικά εγώ υποστήριξα την πρόταση της Επιτροπής για την κατάργηση των οκτώ οδηγιών. Πιστεύω ότι η πρόταση της Επιτροπής είχε σκοπό να απλουστεύσει το ευρωπαϊκό δίκαιο και να εφαρμόσει καλύτερη νομοθεσία δεν ε, επιδιώκουμε την αναρμόνιση πάση θυσία. Πρέπει να σκεφτούμε την εφαρμογή των άλλων οργάνων, ε, των άλλων μέσων και των διεθνών προτύπων αυτά τα εναλλακτικά μέσα πρέπει να εφαρμόζονται εκεί όπου αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική εφαρμογή του. Σχετικά με τη μετρολογία, εγώ είμαι υπέρ της, του εθελοντικού συστήματος αμοιβαία αναγνώρισης με με βάση τα διεθνή πρότυπα. Λυπάμαι που το Κοινοβούλιο μαζί με ορισμένα κράτη-μέλη δεν υποστήριξε αυτή την ελεύθερη και ε, προσέγγιση και προτίμησε μια πιο συντηρητική προσέγγιση. Παρόλα τα αυτά, συγχαίρω τον εισηγητή που αναζήτησε συμβιβαστικέ λύσεις. Εκτιμώ τις προσωπικές του προσπάθειες, χάρη στι οποίε δεν ε, μπήκε στο χρονοτούλαπο αυτό το σχέδιο κειμένου. Ο κύριος Ρώση, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαστε υπέρ αυτή τη έκθεση για τη μετρολογία. Πρόκειται για ιδιαίτερα τεχνικό κείμενο, το οποίο έπρεπε ήδη να είχε ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Δεν προέκυψαν εμπόδια στην ε, αρμόδια επιτροπή. Χρειάστηκε στο Συμβούλιο μεταξύ των 7 κρατών μελών να βρεθεί μια συμφωνία για τους πίνακες συσχέτισης και γι' αυτό καθυστέρησε η όλη υπόθεση. Η Επιτροπή δεν έχει ακόμα υποβάλει την πρότασή της για τα όργανα μέτρησης που θα αντικαταστήσει τα, τις οδηγίες που θέλουμε να καταργήσουμε σήμερα. Εγώ επικρίνω την Επιτροπή διότι προχώρησε σε αυτή την κατάργηση χωρίς να μας υποβάλει την πρόταση αναθεώρησης το, της οδηγίας για τα όργανα μέτρησης. αυτό δεν είναι κάτι που, αυτό που θέλουν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες πολλοί πιστεύουν ότι τα κράτη-μέλη δεν θα μπορέσουν να προσαρμοστούν. Αλλά οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν μάθει να λειτουργούν με τα διεθνή πρότυπα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να φανταζόμαστε ότι θα επέλθει καταστροφή μετά από αυτή την κατάργηση των οδηγιών. Υπάρχει νομοθετικό κενό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι συσσωρεύονται οι κανόνες και είναι υποχρεωμένη να αναζητήσει κανόνες για να εγγυηθεί μια ισορροπία στην αγορά. Παρόλε αυτές τις δυσκολίες, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν μπορούν να λειτουργούν στο, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει να ε, ε, προβάλλουμε υπερβολικές απαιτήσει. Πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνίες μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων πέρα από τις υπάρχουσες πολιτικές διαφορές. Η κυρία Ρόιτοβα, δύο λεπτά η κατάργηση αυτών των οδηγιών δεν είναι σημαντικό πολιτικό ζήτημα. Μιλάμε για την συγκεκριμένη εφαρμογή της αρχής επικουρικότητας και της ανάγκης για καλύτερη νομοθεσία. Υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα διεθνείς συμφωνίες οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την παγκοσμιοποίηση της έρευνας και του εμπορίου. Η εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν απαιτείται οπωσδήποτε. Ε, συμφωνώ με την προσέγγιση της εισηγήτριας που στήριξε την πρόταση της Επιτροπή για την κατάργηση των οδηγιών, ενώ από την άλλη πλευρά για αυτή την οδηγία αφήνει κάποιο χρόνο στις αρχές τις μετρολογικές των κρατών μελών, ώστε να μπορέσουν να προβούν σε μία ανάλυση των επιπτώσεων αυτής της κατάργησης πάνω στην εθνική νομοθεσία. Αυτή η προσπάθεια θα είναι ένα πείραμα ενδιαφέρον και για άλλες οδηγίες, για να δούμε κατά πόσο η αρχή της αμοιβέ αναγνώρισης αρκεί για να μην υπάρξει νομική αβεβαιότητα. Πράγματι, με εκπλήσει το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη προτιμούν την εναρμόνιση. Ολοκληρώνοντας, συγχαίρω την εισηγήτρια η οποία εξασφάλισε την πλήρη υποστήριξη της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ και η οποία κατάφερε να βρει και μια συμβαστική λύση με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάρμπορ. Πρόεδρε, καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Βάισμπεργκερ που είναι ένα παλιό και επιμελές μέλος της Επιτροπής μας. Όταν ξεκίνησε να δουλεύει στο θέμα αυτό, λίγο μετά τις εκλογές πέρσι, όλοι θεωρήσαμε ότι μια απατηλά απλή επιτροπή, ε, έκθεση ε, κείμενο της Επιτροπής θα ξεπερνιόταν, θα τελείωνε γρήγορα και χωρίς πολλές συζητήσει. Νομίζω ότι ο χρόνος που πήρε και η περιπλοκότητα της λύσης δείχνει ότι η απορρίθμιση και η μείωση της γραφειοκρατίας δεν είναι καθόλου εύκολη. Είναι εύκολο να έχουμε όλες αυτές τις φράσεις ε, μείωση της νομοθεσίας. Στην πραγματικότητα ωστόσο πάντα υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να κρατήσουν τους νόμους. Όταν έφτασε αυτό στο Συμβούλιο διαπιστώσαμε κάποια από τα βαθιά ριζωμένα προβλήματα σε χώρες που είχαν προβλήματα για την μέτρηση της χωρητικότητας των εξαμένων των σκαφών, τα αλκοολόμετρα. Ο καθένας έχει το δικό του πρόβλημα. Λοιπόν, το συμπέρασμά μου είναι, όχι κατά πόσο είναι πρόταση είναι καλή όχι, ούτως ή άλλως σε, λίγες, σε λίγους μήνες θα έχουμε την εναλλακτική λύση, που θα είναι την, μια νέα λύση που θα είναι ενημερωμένη. Θα μπορούσαμε να είχαμε περιμένει κάτι τέτοιο, αλλά ζητώ από την Επιτροπή να εξετάζει καλύτερα τις προτάσεις αξιολόγησης αντικτύπου πολύ πιο προσεκτικά πριν υποβάλει νέες προτάσεις εν γέννη. Πιστεύω ότι αν είχαμε περισσότερο χρόνο, περισσότερο χρόνο θα είχαμε σταθεί περισσότερο στο θέμα αυτό. Είναι επιτυχία της Επιτροπής, αλλά επιτυχία με κάποιο μέτρο και πρέπει να μάθουμε τα μαθήματα από αυτά. Ο κύριο Κέλλη στη διαδικασία Catch the Eye. Έχετε το λόγο. Και εγώ καλωσορίζω την πρόταση. Όντως ζούμε σε έναν κόσμο πιο μικρό. Η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων μεγαλώνει και αυτό θα αυξηθεί περισσότερο στο μέλλον. Όσο καλύτερη εναρμόνιση των οργάνων μέτρησης, τόσο καλύτερα. Καλωσορίζω λοιπόν την κατάργηση των οδηγιών για τη μετρολογία και την μείωση κατά 25% της γραφειοκρατίας. Υποτιμώ μερικές φορές τη δυνατότητα των ανθρώπων να προσαρμόζονται. Ο κόσμος προσαρμόζεται πολύ πιο εύκολα. Θυμηθείτε πόσο εύκολα περάσαμε από τα, τις λίρες και τα φαρδίνια στα, ε, στα ευρώ και στα, ε, και στα λεπτά. Από τα μίλια στα χιλιόμετρα. Ήταν εύκολο να είναι, ήταν ευκολότερο από ό,τι νομίζουμε λοιπόν. Πιστεύω ότι η πρόταση αυτή είναι ένα βήμα προ του καυτές μου. Κύριε Πίτρο, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ και όλους τους βουλευτές που μετέσχουν στη συζήτηση γιατί δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον σε αυτή την πρόταση απλοποίηση. Θέλω να υπογραμμίσω εκ νέου τα πλονεκτήματα αυτής της επιλογής και τις θετικές συνέπειες που προκύπτουν. Είναι πλεονεκτήματα υπέρ των καταναλωτών, των παραγωγών ε, εργαλείων και των εθνικών υπηρεσιών. Θέλω να διαβεβαιώσω τους ε, βουλευτές, ιδίως αυτό που είπε η κυρία Γκέπχαρτ, ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε σαν Επιτροπή τα αναγκαία, τις αναγκαίες έρευνες για να προχωρήσουμε σε εναρμόνιση μέχρι τον Απριλίο του 2011. Απαντώντας τώρα στον κύριο Ρώση που έφυγε από την αίθουσα αλλά επέκρινε την Επιτροπή. Καλό είναι να κάνεις κριτική αλλά να ακούς και τις απαντήσεις. Καλό θα ήταν. Υπάρχει κοινή δήλωση Κοινοβουλίου Επιτροπής Συμβουλίου για το θέμα που λέει ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 της Οδηγίας 2004-22 ΕΟΚ ε, για τα όργανα μέτρησης η Επιτροπή καλείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να παραπέμψει, να, να εξετάσει μέχρι τις, το 2011 τις ε, απόψεις για την υλοποίηση της οδηγίας, για την ε, της οδηγίας και να υποβάλει σχετική σε αναθεώρησης. Εγώ, όπως είπα κατά τη διάρκεια της ζήτησης, θα τηρήσω την δήλωση αυτή. Ευχαριστώ τους, ε, ευχαριστώ και εσάς κύριε Πρόεδρε και τους βουλευτές ό,τι αφορά τον πίνακα αντιστοιχίας, αντιστοιχία η Επιτροπή που στηρίζει τη θέση του Κοινοβούλου. Ευχαριστώ. Η κυρία Βάις Γκέρμπερ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την πολύ χρήσιμη συμβολή τους στην απόψινή συζήτηση. Μετά την αυριανή ψηφοφορία θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει από δύο και πέρα. Περιμένουμε τη θέση, την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδηγία για τα όργανα μέτρησης, ώστε να δούμε αν μπορούμε να εντάξουμε τα όργανα στα οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως χωρίς να δημιουργηθεί νομικό κενό. Η κυρία Γκέμπαρτ επέμενε σε αυτό το σημείο το, κάτι στο οποίο, το οποίο μπορούμε να ικανοποιήσουμε. Είμαι βέβαιη και τα κράτη-μέλη καλούνται να αποδείξουν ότι ορισμένα στοιχεία θα υπάρχει δυνατότητα να διατηρηθούν με ανυπομονησία και τις ε, διαβουλεύσεις ε, στο ίντερνετ ε, που έχει εξαγγείλει η Επιτροπή, δηλαδή θα συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείε κλπ. Εγώ θεωρώ ότι όσον αφορά ορισμένα όργανα μέτρησης, για παράδειγμα τα αλκοολόμετρα, ε, έκανα μια σχετική έρευνα ε, και μου είπαν ότι ε, στην πραγματικότητα δεν χρησιμοποιούνται καθόλου πλέον. Και αν θέλουμε να προσεγγίσουμε το στόχο το 2012 να έχουμε μείωση της γραφειοκρατίας στην Ευρώπη θα πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα. Εγώ είμαι διατεθειμένη, μάλλον εμείς ως Κοινοβούλιο είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε τη δική μας συμβολή. Και κλείνοντα θα ήθελα να πω ότι ναι ε, ήταν ένα συμβασμός αλλά θα ήθελα μελλοντικά να καλέσω και τις, τις χώρες μέλη ε, να να εθετήσουν ε, δεσμευτικούς στόχους γιατί πραγματικά είναι σημαντικό να υπάρχει μια ενιαία ρύθμιση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και τον Επίτροπο. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη.